ομιλίες ενός λεπτού βάσει του άρθρου 163. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ιβαν Στέφανετς. pán predsedajúci doprava v mestách sa stáva neustále pálčivejšou témou ktorú je treba riešiť. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα ποδήλατα θέλω να μιλήσω. Η κυκλοφορία στις πόλεις είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Χρειαζόμαστε πολλές διαφορετικές λύσεις. Μία λύση θα ήταν να χρησιμοποιούνται ευρέως τα ποδήλατα. Είναι πιο περιβαλλοντικός φιλικά. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα ποδήλατα μπορούν να προχωρούν πιο γρήγορα από τα αυτοκίνητα, ιδίω στις περιπτώσει συμφόρηση, ώρες αιχμής. Στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε περισσότερους ποδηλατοδρόμους, ιδίως κοντά σε σταθμούς και σε σημεία κομβικά. Εκεί χρειαζόμαστε ποδηλατοδρόμους. Πιστεύω Εδώ πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και ήθελα να πιστήσω την προσοχή σα αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Βίκτορ Νεγκρέσκου από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω για τις σοβαρές διακριτικές ε, μεταχειρήσεις κατά των Ρουμάνων στη, Μέλη ε, μεταξύ των οποίων στην Ιταλία δεν εκπροσωπούνται έτσι όλοι οι Ρουμάνοι με τη ρατσιστική αυτή συμπεριφορά εναντίον τους. Έχουμε πολλές φορές την εντύπωση ότι οι Βρετανοί επίσης έχουν πολύ σοβαρές προκαταλήψεις κατά των Ρουμάνων. Θα ήθελα να υπερασπιστώ τους ε, Ρουμάνους που, ε, που, που κατοικούν στην Ελλοδαπή δεν αντιδρούν οι ευρωπαϊκοί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει κάθε ρατσιστική ξενοφοβική τοποθέτηση, ακόμα και αν πρόκειται ε, για συναδέλφου του Ευρωκοινοβουλίου ή για οποιονδήποτε πολιτικό. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα οργανώσει μια εκστρατεία κατά της διακριτικής μεταχείρισης για να δείξει ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ε, ρατσιστική εκδήλωση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρασνέψκη από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το κοσυφοπέδιο. Πρόσφατα ε, είδαμε ε, νέα κύματα μετανάστευσης ε, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από το κοσμοπέδιο κυρίως προς τη Γερμανία και πολλοί λένε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να ανακόψουμε αυτή τη μετανάστευση. Πραγματικά μας απογοητεύει αυτό το γεγονός. Ασχολούμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο με οτιδήποτε, επί παντός επιστητού, δίνουμε συμβουλές, λέμε σε όλους πώς πρέπει να οργανώνουν την οικονομική, πολιτική του ζωή. Ασχοληθήκαμε και με τη Βενεζουέλα πριν, ενώ δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας. Δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο μεγάλες χώρες όπως η Ουκρανία, ούτε και μικρότερες όπως το Κοσμοπέδιο. Παρά τα 2 δις ευρώ του ε, προπολογισμού που έχουμε δώσει από το παρά το Eurolex, παρά την παρακολούθηση τη κατάσταση στη χώρα. Η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ άσχημη. Για το 2013 ο δείκτης εξαθλίες από το Business Insider βάζει ε, στις 25 χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις στο κοσμοπέδιο, μαζί με το Αφγανιστάν, το Μαλί και το Νότιο Σουδάν. Επομένως είναι δύσκολο να σκεφτούμε ε, γιατί κάποιος θέλει να φύγει από αυτή τη χώρα. Αντί λοιπόν να συζητάμε όλα αυτά τα προβλήματα του υπόλοιπου κόσμου, γιατί να μην συζητήσουμε τα δικά μας προβλήματα. Και ίσως μας ακολουθήσει τότε και ο κόσμος. Ευχαριστώ. Από την άλλη η επόμενη ομιλήτρια, Αγγέλικα Μιντνερ. Θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, διακρίσεις ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, τη διαδικασία που ξεκίνησε από την ε, Αυστριακή ε, Εισαγγελία κατά ενός ατόμου που δημοσίευσε μια φωτογραφία του Χίτλερ και είχε κάποια λεζάντα που ασκούσε κριτική κατά του Ισραήλ. Αυτό όμως ήταν θεμητό. Ουσιαστικά δεν πρόκειτο για στήριξη του ναζισμού. Από το 2008 έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για να εξαλείψει τις διακρίσεις επί τη βάση φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προσέγγισης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ε, πρακτικές και να έχουμε νομοθεσία η οποία θα προστατεύσει τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Χρυσογόνος έχει το λόγο. Από την ΚΟΕ. Ένα λεπτό. Στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ο ελληνικός λαός ψήφισε κατά της συνέχισης της καταστροφικής πολιτικής λιτότητας. Η αποτυχία της πολιτικής αυτής προκύπτει μέσα από τις ομολογίες των ίδιων των εμπνευστών της, όπως η παραδοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για χονδροειδή υποτίμηση του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, δηλαδή των υφεσιακών επιπτώσεων της λιτότητας. η νέα κυβέρνηση έχει εισέλθει σε μια τετράμινη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς του δικού της σχεδίου για την ανασυγκρότηση της χώρας. στο πλαίσιο αυτό η ευρωπαϊκή επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση του ελληνικού λαού και να αποδεχθούν δραστικές αλλαγές στο μείγμα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής οι οποίες απαιτούνται προκειμένου η ελληνική οικονομία και κοινωνία να τεθούν σε βιώσιμη τροχιά. μόνο έτσι μπορεί η ένωση να φανεί συνεπής προς τις αξίες της δημοκρατίας και της επικουρικότητας που περιέχονται στην ιδρυτική της συνθήκη. Ευχαριστώ. πολύ. Ο κύριος Ρόπε από την ομάδα των σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, χθες έλαβε χώρα ένα συνέδριο γαλακτοπαραγωγών στην Λιθουανία. Οι παραγωγοί της Λιθουανίας προσπαθούν να βρουν μια λύση στο πρόβλημα του αν χρειάζεται ακόμα κανείς το γάλα τους. Παίρνουν μονάχα 12 σέντ το λίτρο του γάλακτος και αυτό είναι χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής. Οι βαλτικές χώρες δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό αντιστάθμισμα για το ρωσικό εμπάργο, για το εμπάργο κατά της Ρωσίας. Η παραγωγή γάλακτος λοιπόν βρίσκονται σε μια απελπιστική κατάσταση. Είναι γνωστό σε όλους ότι η γαλακτοπαραγωγή της Λιθουανίας παίρνουν πολύ χαμηλές πληρωμές και αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τιμή του γάλακτος είναι πολύ χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής <clears throat> το οποίο αυξά, αυξάνεται συνεχώς την τελευταία δεκαετία. Γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να προστατεύσουν τους γαλακτοπαραγωγούς της Λιθουανίας. Ευχαριστώ. Ο Φάμπιο Μπάσιμο Καστάλδο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους αν ξέρουν τι είναι αυτό. Αυτό είναι φωτογραφία από ε, μια, ένα πανό που από ένα μπλουζάκι μάλλον που εμφανίστηκε στο ίντερνετ μετά από όσα συνέβησαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Ρώμη της περασμένης εβδομάδας με τη Ρώμη Φάγενορντ και είναι ε, μπλουζάκι φιλάθλων. Αυτές, ε, αυτό το όνεδος δεν μπορεί ακόμη να επιτρέπεται. Έχει πολύ σοβαρές ευθύνες, έχουν πολύ σοβαρές ευθύνες οι Ιταλικές αρχές για την διαχείριση αυτής της κρίσης, αλλά εντωμεταξύ καταστράφει ένα άγαλμα και ένα συντριβάνι ανεκτήμητης αξίας πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Ε, και βεβαίω οι ζημιέ που έχουν επιφερθεί είναι αμετάκλητε. Δεν μπορεί λοιπόν το ποδόσφαιρο που είναι άθλημα να έχει τέτοια εξέλιξη. Θα πρέπει και οι συνάδελφοι και εμεί να αναρωτηθούμε τι γίνεται και μαζί με του συναδέλφου να φέρουμε το ποδόσφαιρο στο πραγματικό του ύψο. Δεν μπορεί να προξενεί βία, ούτε να επιτρέπουμε τη βία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε. Κυρία Ντότς. μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την ευκαιρία να εκφράσω τις ειλικρινείς ανησυχίες των ε, ψηφοφόρων μου από τη Βόρεια Ιρλανδία για το Ταμείο ε, Κοινωνικής ε, Στήριξης. Υπάρχει ένα μέρος πολιτών που πιστεύουν ότι έχουν τύχει μη διαφανούς και άδικες μεταχειρήσεις από τις αρμόδιες αρχές. στο πρώτο στάδιο της αίτησής τους, 60% ποσοστό αποτυχίας διαπιστώθηκε και 12 τουλάχιστον μάλλον 100 ε, άνθρωποι ειδοποιήθηκαν για, για την πρόθεση να απολυθούν και πολλές θέσεις μαθητές ασκουμένων πρόκειται να καταργηθούν. Εδώ λοιπόν αυτό ε, αφορά ολόκληρα σοβαρά ε, μεγάλα, μεγάλες ομάδες της κοινωνίας μας. Υπάρχει κοινωνική ένταση, θα σας ζητούσα να να ερευνήσετε το τι γίνεται με την περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας και βάσει του κανονισμού με τις κοινέ διατάξεις που ορίζει ότι η επιλογή των προγραμμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις και με τρόπο διαφανή. Έκλεισε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το 30% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τη Βόρεια Ιρλανδία να ε, στοχεύει όντω την εκρίζωση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ε, συμπερίληψης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γολάν. Οι χαλιβουργικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ζουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενώ ο χάλιβας είναι πάρα πολύ σημαντικός σε πολλές παραγωγικές διαδικασίες και ο ανοξίδωτος χάλιβας αντιμετωπίζει αθέμητες πρακτικές και το dumping που ασκείται από τη Κίνα. Για τους εργαζόμενους στην ε, ε, στο Βέλιο υπάρχουν τρομερά προβλήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αθέμητες πρακτικές που καταστρέφουν τη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλήρως τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Είναι απαραίτητο το ταχύτερο δυνατό να συνεδριάσει η ομάδα υψηλού επίπεδου για το χάλιβα και να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική στρατηγική που θα δώσει ένα μέλλον στην χαλιβουργία μας και ιδίως στον ανοξίδωτο χάλιβα η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις, αλλά χρειάζεται και πραγματική υποστήριξη στη βιομηχανία μας. Θα πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας την ικανότητα να μπορούμε να αποφασίζουμε σύντομα και αποφασιστικά. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί. Η κυρία Τζοφρίντα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ήθελα για άλλη μια φορά να αναφέρω στους συναδέλφους το θέμα της μετανάστευσης της 2 ε, Οκτωβρίου 2013 ήταν, είναι μια μέρα θρήνου για την, και πένθους για την ε, Λαμπεντούζα που άφησε άφωνο τον κόσμο ε, και 15 μέρες πριν μόλι, μόλις είχαμε άλλους 300 νεκρούς που θα βαραίνουν τις συνηθίσεις μας. Ενώ τα μέσα μαζική ενημέρωση όλου του κόσμου λένε ότι η Ευρώπη απλώ κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έτσι ε, όντω η Ευρώπη καθυστερεί. Τι περιμένουμε, η Μέση Ανατολή είναι αποθήκη. η Βόρεια Αφρική ε, είναι ανεξέλεγκτη. Οι περιοχέ σύγκρουση και εστί πολέμου ε, σπρώχνουν εκατομμύρια άντρε και γυναίκε να βγουν στη θάλασσα και να αναζητήσουν διέξοδο. Ε, είναι τεράστιος ο αριθμός των θανάτων. Φτάνουν τα λόγια, φτάνει η σιωπή. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος και μια ε, πολιτική κατανομή των ποσοστώσεων, ώστε όλοι τα κράτη-μέλη, χωρίς καμία εξαίρεση, να αναλάβουν την ευθύνη για αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φωτίνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Κέντρο Αριστείας της Ρήγας για το ΝΑΤΟ ετοίμασε μία μελέτη για την προπαγάνδα της Ρωσίας, την προπαγάνδα που προηγήθηκε της επίθεσης κατά της Ουκρανίας και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων αυτών. Στην μελέτη αυτή εντοπίζεται πώς ο ελεύθερος κόσμος παραπληροφορήθηκε για το τι ε, πραγματικά συνέβαινε στην Ουκρανία. Επίσης, σημαντικό είναι το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δημοκρατικές χώρες προσκαλούν τις ρωσικές αρχές στον Μπρισμπέιν, στο Μόναχο και τον ε, Πούτιν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Ίσως δεν καταλαβαίνουμε ότι μας ε, ε, χρησιμοποιούν για την, για την προπαγανδιστική τους μηχανή οι Ρώσοι διότι τους επιτρέπουμε να έχουν μια θέση από την οποία μπορούν να ενεργήσουν. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ρωσία είναι ένα κράτος που είναι επιθετικό στις δράσεις του κατά άλλων ε, κυρίαρχων χωρών και θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε στηρίξη σε αυτού του είδους της δράσης και της ανάγκης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάτ Μακάρθη από την QNGL. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το TTIP θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη διμερή εμπορική συμφωνία στην ιστορία. Οι πολίτε όμω τη Ευρώπη ε, αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανησυχία ε, την όλη διαδικασία και αμφισβητούν και για την, ακεραιότητα και για την ακαιρεότητα της Κομισιόν. Για μένα είναι πάρα πολύ πρόωρο. Ε, θα πρέπει να είχε υπάρξει συζήτηση πριν καταλήξει η Ευρώπη στις θέσεις της. Όμως η Κομισιόν δεν το έκανε και πολύ κρυφά ε, συνέχισε μέχρι πρόσφατα τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε το μηχανισμό ISDS ε, που θα δίνει δυνατότητα σε εταιρείε να απειλούν εκλεγμένες κυβερνήσεις και να παραγνωρίζουν ε, το κράτος δικαίου, την εγχώρια νομοθεσία. Αυτό είναι κάτι που βρίσκει τεράστια αντίσταση. Εμείς επίσης δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, άνοιγμα περαιτέρω των αγορών μας, μείωση των τιμών, ούτε ε, να ε, υποβαθμιστούν τα πρότυπα και να μπούμε σε μειονεκτική θέση ως αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει η Κομισιόν ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα πρότυπα. Δεν έχουμε δει ακόμη όμως προτάσεις που να μας πείθουν για το τι θα συμβεί αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα κέρδη θα είναι πολύ μικρά σε σχέση με τις τεράστιες απώλειες που θα έχουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εταιρεία Κροαζιέρες Κώστα μετέφερε ε, εκατοντάδες εργαζομένους από την Γένοβα στο Αμβούργο χωρίς να ε, συνεννοηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους και από μετά από μια σειρά δηλώσεις εκφοβισμού και προσβλητικές προς τους εργαζομένους από την πλευρά των αρχών της εταιρείας. Αναρωτιέμαι αν αυτή η συμπεριφορά μπορεί να γίνεται δεκτή και να μην θεωρείται και παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας και της ε, ευρωπαϊκής. Θα πρέπει, ακόμη και αν δεν είναι έτσι, να τονίσω ότι πρόκειται για όνειδος. Είναι ντροπή να μην που δεν υπάρχει και δεν δικαιολογείται από κανένα οικονομικό λόγο για την μετατόπιση των εργαζομένων αυτών και μια ε, εταιρεία ε, που ε, έχει την βασική της δύναμη στην Ιταλία και θέλει και εκμεταλλεύεται εκατοντάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ εκ μέρους της Ιταλίας υλικά μετατοπίζει του εργαζόμενου σε άλλες χώρες, τις θέσεις εργασίας σε άλλε χώρε, Μιλάμε για πόλει τουλάχιστον για 300 άτομα και για απώλεια θέσει τουλάχιστον 60 θέσεων εργασία. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη την οποία ονειρεύομαι κύριε Πρόεδρε και δεν είναι δίκαιο κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μπούντα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης είναι και μια εγγύηση για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και του επίπεδου απασχόλησης των πολιτών μας. Το σχέδιο επένδυσης ε, Juncker εκπροσωπεί 315 δισεκατομμύρια ευρώ και επίσης το πρόγραμμα Horizon 2020 και το πρόγραμμα Erasmus και τα κονδύλια της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι οι κύριοι άξονες χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη. <clears throat> Πολλά όμως κράτη-μέλη έχουν πραγματικές δυσκολίες για να μπορέσουν να απορροφήσουν τα κονδύλια αυτά λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών τους. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν και το Συμβουλίο να απλοποιήσουν αυτές τις διαδικασίες και να εξασφαλίσουν την ε, ενοποίησή τους για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε η, τα ταμεία συνοχής και τα διαφορετικά ταμεία να γίνουν πραγματικότητα για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τανσέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι η διατλαντική εταιρική σχέση για το εμπόριο και τις επενδύσεις, TTIP, είναι μια εμπορική συμφωνία που μπορεί να φέρει σημαντικούς, σημαντικά ωφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Τα προβλήματα των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνουν στο μυαλό μας όταν συζητούμε και διαπραγματευόμαστε αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να υπονομεύσει την κατάσταση των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ήδη ε, αρνητική και να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου οι Ευρωπαίοι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν ακόμα περισσότερο για τα νέα φάρμακα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να δρούν με τρόπο διαφανή και να θέτουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών τους για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Θα πρέπει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπονομευτεί η αρμοδιότητά της στα θέματα των φαρμακευτικών προϊόντων. Δεν πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα στα κράτη-μέλη και να περιοριστεί η δυνατότητα δράση εναντίον των φαρμακευτικών εταιριών. Το πιο σημαντικό προέχει είναι η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φων Στόρχ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ισλαμικό κράτος σκότωσε 11 άτομα τα οποία αποκεφάλισε στη Λιβύη πριν από μερικές μέρες. Είναι μια αιματηρή ιστορία η οποία στρέφεται κατά των κρατών των σταυροφοριών, όπως λένε. Θεώρησε το Ισλαμικό καθεστώς ότι έπρεπε να σκοτώσει τα άτομα αυτά επειδή είναι χριστιανοί. Αλλά δεν σκοτώνουμε χριστιανούς στο Ισλαμικό κράτος δεν σκότωσε μονάχα 21 χριστιανούς, αλλά και 21 ομοφιλόφιλους. Αυτό ακριβώς συνέβη. Θα έπρεπε κανείς να περιμένει να υπάρξει η αλληλεγγύη και η υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αλλά δεν ακούστηκε καμία κραυγή αγανάκτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσατε μονάχα ότι σκοτώθηκαν χριστιανοί. Τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο Πολ Τσακί από το ΕΛΚ, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από 9 χρόνια, το 2006, άγνωστοι επιτέθηκαν σε μια ε, Ουγγαρέζα ε, φοιτήτρια γιατί χρησιμοποίησε τη μητρική τη γλώσσα. Τότε ο Υπουργός Εσωτερικών είχε πει ότι θέλησε να πλήξει ε, την ε, φήμη της Σλοβακίας. Ε, η κοπέλα που ήταν επινόησή της σε όλη η ιστορία. Έξι χρόνια λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία η κυβέρνηση τελικά ζήτησε συγγνώμη στο κορίτσι αυτό το οποίο στο μεταξύ είχε καταφύγει, είχε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ξαναξεκινά όμως αυτή η διαδικασία. Και η φοιτήτρια αυτή που έφυγε από τη χώρα και διαμένει σε άλλο, ε, έχει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω αυτής της δίκης που θα ξαναγίνει όπου να είναι και θα πρέπει να παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ, Αλφρετ Σάντε. Τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πριν από λίγα χρόνια θέλαμε ένα σύνταγμα για την Ευρώπη και υπήρχε και συντακτική συνέλευση, αλλά ε, το απέρριψαν οι ευρωπαϊκέ χώρε και ήταν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μεταξύ είχε δημιουργηθεί η Νομασμοτική Ένωση, χωρί να υπάρχει η απαραίτητη οικονομική ένωση, με μεγάλε αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωζώνη γνωρίζει ύφεση, με ευάλωτε υποδομέ από ό,τι φάνηκε. Αλλαγέ προβλέφθηκαν για να αντιμετωπιστεί αυτό σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, όμω με την Νομασματική Ένωση Τελικά δεν έχουμε ένα κεντρικό δημοσιονομικό μηχανισμό. Οι ανισορροπίε και οι ανισότητες ε, τελικά ε, μεταξύ περιφέρειας και κέντρου ουσιαστικά επιβάλλουν πίεση από το κέντρο προς την περιφέρεια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να σώσει την Νομισματική Ένωση από την παράλυση, αλλά ε, δεν το κατάφερε αυτό διότι η Νομισματική Ένωση ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί με τους μη εκλεγμένους εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας να απαιτούν ε, λιτότητα. Πολλοί από εμά πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι απλώς μια θεωρία και θεωρούν ότι η οικονομική διακυβέρνηση δεν προχωρά όπως πρέπει. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε όσα ζητούν οι λαοί και να υπάρχει ε, οικονομική ένωση μεταξύ ε, κυρίαρχων ε, κρατών ή ομοσπονδιακή δομή. Ευχαριστούμε κύριο Σουγιαντόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να μιλήσω για το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών. Ένα νέο δικαίωμα που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και συγκεκριμένα για το πώς ε, εφαρμόζεται, διότι δυστυχώς υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ ε, μεταξύ μας, ε, μεταξύ των πολιτών μάλλον, είδαμε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια να απαιτούν νομική δράση με τις υπογραφές τους για την προστασία των αγέννητων των βρεφών μάλλον, των αγέννητων βρεφών, ε, των εμβρίων. Ο Επίτροπο Τίμερμαν ε, δηλώνει τώρα ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν ε, πρέπει να τύχει νομική μεταχείριση, αλλά πολιτικής. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα γίνει. Αύριο θα υπάρξει δημόσια ακρόαση για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Σα απευθύνω έκκληση να βεβαιωθούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή εξασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών μας και ότι δεν παραμένει κενό γράμμα επί χάρτου. Σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Κλούν από το ΕΛΚ. Η κυρία Κλούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο όλες οι κυβερνήσεις <clears throat> να βοηθήσουν την πραγματική οικονομία με το να υπάρξει ανακαίνιση των δημοσίων και ιδιωτικών κτίριων για να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει πάρα πολλά χρήματα από την ε, ανυπαρξία της ε, μόνωσης. Αυτό μπορεί να δώσει πολλά εκατομμύρια, 450 ευρώ ανα, ανακατοικία με τον τρόπο αυτό. Μπορεί έτσι να καλυφθεί ε, το κόστος της ενέργειας το οποίο χάνεται σε αυτά τα κτίρια. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στην ε, Ιλανδία που συνολικά κοστίζουν πάνω από 600 εκατομμύρια το χρόνο σε φωτισμό και θέρμανση. Με την διαδικασία αυτή θα βοηθήσουμε την απασχόληση, θα βοηθήσουμε τις αγροτικές περιοχές μας, θα ανακάμψει ο τομέας ενέργειας και θα μπορέσει να προωθηθεί και το σχέδιο δράσης του κυρίου Γιούνκερ για να υπάρξει ιδιαίτερα εστίαση στις ε, ενεργειακή εξοικονόμηση στα σπίτια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Τσάμπα Μόλτερ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Ούγγρος ε, Πρωθυπουργός, η ε, Ούγγρική Κυβέρνηση τέλος πάντων, δέχεται κριτική. Τότε οι βουλευτέ του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε λένε ότι η Ουγγρική κυβέρνηση κέρδισε δημοκρατικέ εκλογέ, πήρε την υποψία των δύο τρίτων λόγω ε, τη σχετική το θέλησε ο Ουγγρικό λαό. Δεν ισχύει όμω αυτό, διότι ο ΑΣΕ είπε ότι η πλειοψηφία των δύο τρίτων επετεύχθη λόγω αλλαγών του εκλογικού συστήματος και της παρουσίας ε, ε, αυτού των εκπροσώπων του κόμματος στον τύπο και στα μίντια. Αρνητικό δηλαδή, αρνητική τιμιγορία για την ε, εγκυρότητα των εκλογών. Την Κυριακή, στο Βέστριμ, εξέφρασε ο λαός τη βούλησή του όπου σε μια εκλογή που έγινε παράπλευρη ε, κέρδισε αντιπολίτευση. Και αυτό τελειώνει με την πλειοψηφία των ε, δύο τρίτων την κυβέρνηση. Έτσι μπορούμε πια να ξαναμπούμε στο δημοκρατικό μονοπάτι. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Μαριάννα Πετήρ. Πιστεύω στο κράτος δικαίου και θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να τηρεί αυτή την αρχή σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις υποψήφιες χώρες. Περιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από τη Σερβία να ακυρώσει τα άρθρα 2 και 3 του νόμου της για, την διανομή, για τη διαμονή και την αρμοδιότητα των κρατικών αρχών για τα εγκλήματα πολέμου, κάτι το οποίο έχει τύχει κατάχρησης από τη Σερβία που δεν δέχεται την αρχή της ε, ε, οικουμενικής δικαιοδοσίας. Παίζει το ρόλο μικρού διεθνούς δικαστηρίου η Σερβία με νομικά κατασκευάσματα που μπορεί να ε, εμποδίσει την είσοδο σε προερχόμενους από 17 χώρες πολίτες που έχουν πολεμήσει στον πολεμό με την Κροατία. Επίσης, είναι σαφές από το ε, από τον πόλεμο του 1991-1995 ότι υπάρχουν καταγγελίες κατά της Σερβίας για, τη διάρκεια, για κλίματα πολέμου. Δεν μπορεί μια τέτοια χώρα όμως να θέτει τους Κροάτες σε δικαστήρια για ενέργειες που έχουν γίνει στο εδαφός. Θα πρέπει να συνεχίσει τον ευρωπαϊκό δρόμο της Σερβία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή την πορεία και να διατηρήσει το κράτος δικαίου, κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε κυρία Μπιγιάννα Μπορζάν από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο εμβολιασμό είναι μια από τα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Για την δημόσια υγεία, οι χώρες επενδύουν ε, στον εμβολιασμό, όχι όμως αυτές ε, του τρίτου κόσμου όπως λέγεται και δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες τους να εμβολιαστούν. Έτσι φτάσαμε το 2013 31.000 θανάτους λόγω έλλειψης εμβολιασμού. Στη Γερμανία, μια από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, πέθανε ένα βρέφος από ασθένεια που θεωρείταν ε, υποέλεγχο. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε την υγεία των πολιτών παγκοσμίω. Αυτοί που να εμβολιαστούν είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της πολιτικής. Εγώ είμαι από την Κροατία, μια χώρα που ε, δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό των παιδιών. Ε, είναι Πολύ σημαντικό όμως ή τα βακτηρίδια και τα μικρόβια να αντιμετωπίζονται όπως πρέπει και είναι, να είναι ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες ως την υγεία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το μέτρο της άρνησης συμβολισμού των παιδιών. Ευχαριστούμε κυρία Αγγέλα Βαλίνα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για την υπατήτη C, που δεν είναι μόνο ένα από τα μεγάλα προβλήματα υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι και το βασικό αίτιο μεταμοσχεύσεων ύπατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχει το Solvay, ένα φάρμακο με 90% επιτυχίας, ε, όπως λέει και η πλατφόρμα των πληγέντων και θα μπορούσε να το αγοράσει κανεί για 100 ευρώ ε, ε, γενώσιμο, αλλά 25.000 ε, το πουλάει η εταιρεία. 4.000 άτομα έχασαν τη ζωή του στην Ισπανία γιατί δεν ε, έδρασε η κυβέρνηση τη Ισπανία. Όπω είχε ορίσει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και είχε εγκρίνει, δεν αγόρασε αυτά τα φάρμακα, τα γενώσιμα, αλλά δίνουμε 11 δις το χρόνο στην Εκκλησία της Ισπανίας. Παραβιάζει οδηγίες η Ισπανία που εγγυώνται το δικαίωμα της προστασίας της υγείας. Ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνα για να δει κατά πόσο πράγματι ε, και ο κανόνας ανταγωνισμού και περί δημοσίων συμβάσεων καταπατώνται λόγω της πολύ ψηλής τιμής των φαρμάκων αυτών. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι ένα άλλο μέτρο που θα μπορούσε να ληφθεί είναι σε περίπτωση που έχουμε καταχρηστική τιμή ε, που επηρεάζει και την ε, βιωσιμότητα να λαμβάνονται μετά. Και παρακαλώ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρίες και η επίθεση του Ισλαμιστικού κράτους οδήγησε και σε άλλη μια φρικαλαιότητα, την θανάτωση 21 χριστιανών της Λιβύης. Οι τζιχαντιστές εμφανίστηκαν στην πόρτα μας, ε, στη Λιβύη και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την άμεση απειλή πλέον. Ε, πέρασα πέντε μέρες σε καταβλισμούς προσφύγων και ήθελα να ευαισθητοποιήσω τις αρχές για τις ανάγκες των πολιτών. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς, ενώ ε, οι ε, προαιώνια χριστιανική παράδοση στη Μέση Ανατολή αφανίζεται. Πρέπει να προστατεύσουμε τι μειονότητε, είτε είναι χριστιανικέ είτε άλλε προέλευσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στο Κοινοβούλιο ζητώντα ε, την ε, να αναλάβει δράση σε ανθρωπιστικά ζητήματα. Ε, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία θα έπρεπε να εξαρκούν για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ιδίως στις χώρες όπου βρίσκονται, για να παραμείνουμε ε, αν παραμείνουμε παθητικοί, ουσιαστικά αντιφάσκουμε με τις αρχές της Ευρώπης και είμαστε απάνθρωποι. Θέλω να καμαρώνω και επιτρέψτε μου να είμαι περήφανος για όσο μπορεί να πετύχει η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τόκες δεν είναι εδώ. Η κυρία Νίνα Γκίλ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τους στόχους του, της Ευρώπης 2020. Μια ευφυά e ε, καινοτόμα μορφή ανάπτυξης. Αλλά ακόμα έχουμε τα ερήπια της κρίσης του 2008. Στα δυτικά Midlands έχουμε μια μεγάλη ανεργία και είναι η τρίτη μεγαλύτερη περιοχή ε, εξαγωγικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και όπου ελείπουν οι απαραίτητες δεξιότητες παρόλα αυτά. Πώς θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη και παραγωγικότητα αν δεν αντιμετωπίσουμε τα τοπικά προβλήματα αυτά χρειαζόμαστε περισσότερο έλεγχο σε τοπικό επίπεδο και λιγότερη παρέμβαση του Λενδίνου. Αλλά ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ζητά κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, υποστήριξη η περιοχή μου έχει την τεχνολογία και το δυναμισμό που μπορεί να κάνουν πραγματικότητα την ανάπτυξη. Οι οικονομίε μα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν μεγαλύτερη επανεξισορρόπηση εξουσιών μεταξύ τοπικών αρχών και εθνικών κυβερνήσεων. Στα κάτι μέρη και για ένα δευτερολεπτάκι μονάχα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να συμμετέχουν οι πόλεις και οι περιοχέ στην διαμόρφωση πολιτικής για να έχουμε προσθέμενη αξία που θα δει και ο ο απλό ο εκλογέας. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα ιδιαίτερα ανεκτικός. Η Μαρίζα Ματίας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Οι τελευταίες εβδομάδες διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση έδειξαν ότι τα προγράμματα λιτότητος ε, δεν λειτουργούν αντίθετα με αυτά που είπαν οι διάφοροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και η πορτογαλική κυβέρνηση. Έχει πέσει 63% το επίπεδο επενδύσεων. Χάθηκαν 220.000 θέσεις εργασίας στην Πορτογαλία και το μόνο πράγμα το οποίο μειώθηκε ήταν το εθνικό χρέος. Ενώ αυξήθηκε η ανεργία και η ένδια. Τον έχουμε ως υπόδειγμα και η ιστορία επιτυχίας στην Πορτογαλία είναι απόλυτα λανθασμένο. Εάν υπήρχε αυτή η κατάσταση δεν θα είχαμε την σημερινή κατάσταση όπου η Κομισιόν θα θέσει υπό την Πορτογαλία για υπερβολικά ελλείμματα. Δυστυχώ είναι ένα παράδειγμα όχι επιτυχίας αλλά αποτυχίας των πολιτικών αυτών η Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ Λέω Πρόεδρος. Ο κύριος Φραντς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Νέε θέσει απασχόληση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην απόγνωση των σημερινών νέων. Ακούσαμε υποσχέσεις ε, ε, που είναι κατά της ε, λογικής, της οικονομικής. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέα απογοήτευση τον κόσμο. Άρα πρέπει να έχουμε μια νομισματική πολιτική ενεργητική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε και το σχέδιο των επενδύσεων, Juncker. Αυτά μας αφήνουν να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια στροφή στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι πολίτες μας χρειάζονται μια τομή. Χρειάζεται μια αλλαγή στην οικονομική πολιτική κατάσταση και ζωή. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε θα απογοητευτούν εκ νέου. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσά, αγαπητέ συνάδελφοι, αλλά και του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να εγκρίνετε το στομότερο δυνατό τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέψουν ε, στα κράτη-μέλη να οδηγηθούν σε οικονομική ανάπτυξη. Ο κύριος Λάσλο Τόκες, ο επόμενος μιλητής. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τα θέματα του κομμουνισμού ήθελα να μιλήσω για την υπόθεση της ε, στην ε, Τη υπερδνηστερίας στη Ρουμανία, όπου η ουγγρική μειονότητα ε, γνωρίζει μεγάλη καταπίεση. Ε, μεταξύ άλλων, έχουμε προχωρήσει πολύ στη Ρουμανία, έχουμε ρίξει τη δικτατορία, αλλά πολύ μεγάλο μέλος του κοινού ε, επιμένει στην ίδια πολιτική του Τσαουσέσκου και υπάρχει ε, τάση απόσχησης της υπερδυνιστερίας με πρόσχημα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προστασία της ουγγρικής μειονότητας. Μιλάμε για σοβαρές ε, παραβιάσεις των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπίεση της ελευθερίας λόγου και της ελευθερίας της συνέχισης. κάτι που ουσιαστικά προστατεύεται από το Ρουμανικό Σύνταγμα. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει υπέρ της περιοχής αυτής και της αυτονομίας της. Σας ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Ήσασταν ο τελευταίος και λουκούμιος ομιλητής στην σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους